Okay, dear colleagues. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της συνεδρίασης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση αυτής. Θα ήθελα να προτείνω να προσθέσουμε κάτι μετά το σημείο 15. Ψηφοφορία για την προσωρινή συμφωνία που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις της, για τα αυτόνομα μέτρα εμπορίου. Αποτέλεσμα της, ε, της συνεδριάσεων περασμένης εβδομάδας στο Στραμσβούργο. Εάν δεν υπάρχει κάποια άλλη επιθυμία να προσταθεί κάτι στα διάφορα, μπορούμε να εγκρίνουμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών. Όπως συνήθως τα πρακτικά εγκρίνονται εκτός αν υπάρχουν αντιρρήσεις ή μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Σημείο 4. Ανακοινώσεις του Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Οι συντονιστές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 3ης Μαΐου. Έχουν λάβει αποφάσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά της συνεδρίασης. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν κάποιες ενστάσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα εγκριθούν και αυτά. Μετά, σημείο 5. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Πρώτα, βλέπετε στα δεξιά μου ένα πρόσωπο από τα παλιά, ο Μάτι Κάραους, ο οποίος διορίστηκε τμήματάρχης και θα είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση της γραμματείας της Επιτροπής μας. Θα θέλαμε λοιπόν να σε καλωσορίσουμε και να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια. So I say... Καλώς όρισες λοιπόν και πάλι στην Επιτροπή μας. Νομίζω πέντε χρόνια εργάστηκε στην Κομισιόν. Όχι, δύο χρόνια, μόνο δύο χρόνια. Μα έλειψε λοιπόν. Τα δύο χρόνια ήταν αιώνε. Νομίζω τώρα έπραξες καλώ και ήρθες με το μέρο του Κοινοβουλίου. Και επίση με το μέρο του Κοινοβουλίου είναι και ο Χέκη, ο οποίος είχε καθήκοντα τμήματάρχη για έξι μήνε περίπου. Ναι. Και εκτέλεσε τα καθήκοντά του εξαιρετικά. Θα ήθελα λοιπόν να τον ευχαριστήσω για τη δουλειά που έκανε τους τελευταίους μήνες. Εκτιμούμε πάρα πολύ τη δουλειά σου. Μετά. Περνάμε σε Άλλες ανακοινώσεις. Στις 31 Μαΐου είχαμε ένα γεύμα για την Συμφωνία TPC. Συζητήσαμε αρκετά θέματα που αφορούν τις εργασίες μας, ιδιαίτερα για τις εμπορικές προτιμήσεις για την Ουκρανία, το Υπουργικό Συνέδριο στα πλαίσια του ΠΟΕ, όπου ζήτησα μια σαφή δέσμευση βασισμένη στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σιγκαπούρης. Δεν έλαβα όμως απάντηση από τα κράτη-μέλη, τα οποία βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία προβληματισμού. Ελπίζω όμως να έρθουμε σε έναν συμβιβασμό για τη δέσμη μέτρων ε, για το εμπόριο και τον εξυγχρονισμό αυτών. Ελπίζουμε να ε, έχουμε αποτελέσματα κατά τη... πριν το τέλος της Μαλτέζικης Προεδρίας, θα δούμε. Και τέλος, είπα ξεκάθαρα ότι είμαστε απογοητευμένοι από την αργή πρώτα των διαπραγματεύσεων για την διαδικασία καλύτερης νομοθεσίας και για την εξωτερική της διάσταση. Το Συμβούλιο δεν προχωρά Και ανέφερα σαφώς ότι αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε μια συμφωνία για την πρόσβαση στα έγγραφα, για την ισότητα στην πληροφορία κτλ., τότε δυστυχώς το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ελπίζω όμως να καταφέρουμε να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό έτσι ώστε να το αποφύγουμε. Τρίτον, αν γνωρίζετε, ο κύριος Ρόμπερτ Λάιτχάιζερ έχει αναλάβει τα καθήκοντά του στην ε, κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Του έστειλα μία συγχαρητήριο επιστολή και τον κάλεσα να έρθει στην Επιτροπή μας ακριβώς για να συζητήσουμε το Υπουργικό Συνέδριο του ΠΟΕ στον Πουένος Άιρες. Αυτά λοιπόν ε, ως προς τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Θα περάσουμε λοιπόν στο σημείο 6 κατάσταση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου. Α, ο κύριος ε, Μόζε είναι εδώ, θα μας τα πει αυτός. Ναι, ναι, ναι, εδώ είμαι, κρυβόμουν. Δεν ξέρω γιατί δεν με βλέπατε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο τριμερής διάλογος για τη Μολδαβία. Είχαμε μία σημαντική νίκη και το λέω αυτό έτσι με μετρημένα λόγια. Φτάσαμε πολύ κοντά στις ε, δικές μας επιθυμίες. Στην ουσία δηλαδή συμφωνήσαμε για την οικονομική διάσταση του πακέτου βοήθειας 100 εκατομμύρια που ε, θα είναι τα μισά σε μορφή δανείου, τα μισά ε, σε μορφή επιχορήγησης. Αυτά υπό οικονομικές και πολιτικές προϋποθέσεις. Θέλουμε η βοήθειά μας να έχει οριζόντιο όφελο στην Μολδαβία. Επίσης δέχτηκε το Συμβούλιο μια κοινή δήλωση η οποία αφορά τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου ως προϋπόθεση για το πακέτο βοήθειας και αυτό θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα θεσμικά της όργανα, ιδιαίτερα στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Κομισιόν, να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις ε, της αλλαγής του εκλογικού συστήματος στη Μολδαβία και το πώς αυτό θα επηρεάσει το κράτος δικαίου, ε, δεδομένης μάλιστα της ε, γνωμοδότησης της Επιτροπής της Βενετίας γι' αυτό. Επίσης, δεχτήκαμε και κάτι πολύ σημαντικό για το Συμβούλιο, για εμάς όχι και τόσο. Να προσθέσουμε δηλαδή κάτι για την καλή διακυβέρνηση. Αυτό ήταν συμβατό με αυτά που είχαμε ήδη συμφωνήσει για το κείμενο, διότι έχει άμεση επίπτωση στο, στην λειτουργία της διακυβέρνησης στη Μολδαβία. Είμαστε λοιπόν αρκετά ικανοποιημένοι με αυτό. Αυτό από πλευρά απαιτήσεων των άλλων θεσμικών οργάνων. Εμεί σε γενικέ γραμμέ ε, Είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχει και η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για τα κονδύλια που έχουν δαπανηθεί στη Μολδαβία τα τελευταία δέκα χρόνια. Αναφέρθηκε η αιρεσιμότητα των τριών δόσεων, της βοήθειας. Όλα αυτά λοιπόν, ό,τι έχουμε συζητήσει σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, ε, καταφέραμε να ε, τα συμπεριλάβουμε στις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Ε, νομίζω πως το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερο συνεχιζόμενος τριμερής διάλογος, προσωρινά ε, περιοριστικά μέτρα για την Ουκρανία και εδώ είχαμε αποτέλεσμα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Βαλέσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρούμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία ότι καταφέραμε να περάσουμε τις ιδέες μας για διάφορα θέματα όπως ε, οι κανόνες για, τις, ε, για την προέλευση, ε, διαδικασίες ανάκλησης, κλίδες ασφαλείας, συμφωνία σύνδεσης και η εξολόγηση αντικτύπου αλλά και η υποβολή εκθέσεων. Το Κοινοβούλιο έχει πολύ σταθερή θέση σε όλα αυτά τα ζητήματα και τώρα η πρότασή μας φαίνεται λίγο πολύ ότι θα συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο. Οι βασικές αλλαγές πέραν της εντολής που είχαμε, ε, βρίσκονται στα παραρτήματα. Όπως ε, Ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να εξαιρέσει την, ε, τις επεξεργασμένες ντομάτες. Τώρα είναι, έχουμε 3.000 τόνους που μπαίνουν πάλι μέσα στην πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε 5.000 τόνους, οπότε βρεθήκαμε κάπου στη μέση. Επίσης, το Κοινοβούλιο ήθελε να εξαιρέσει το το σιτάρι είχαμε 65.000 τόνους, η αρχική πρώτη κομισιόν ήταν 10.000 τόνοι. Θέλαμε να εξαιρέσουμε την α, ουρία που παράγεται στα, α, σε λιπαντικές ουσίες. Όλες οι γραμμές παραγωγής ε, για τον ιουρικό τομέα επανήλθαν, επανεσυχθήσαν στο κείμενο, αλλά οι προτάσεις που έγιναν ήταν ε, ε, έτσι καλολογικές. Το, ε, το μέλι, το καλαμπόκι και άλλα επανησύχθησαν στην πρόταση. Έχουμε λοιπόν τώρα συνολικά την πρότασή μας για τον τριμερή διάλογο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, αλλά υπάρχει και κάτι που μας ενόχλησε κύριε Πρόεδρε και πρέπει να το πω κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι ξεπεράσατε τι ε, αρμοδιότητε που σα είχαν αποδοθεί κάποιε φορέ. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάμε μία φωνή. Η φωνή του διαπραγματευτού είναι αυτή. Το Νομίζω ότι προσπαθήσατε να πάρετε λίγο τα ενία στις διαπραγματεύσεις και προσπαθήσατε να παρουσιάσετε την θέση του Κοινοβουλίου κάποιες φορές σαν να μην ήμουν εγώ παρόν. Και αυτό πραγματικά με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε στο μέλλον αυτό να το επιλύσουμε. Αλλά την Τρίτη όταν διαπραγματευόμασταν ε, εκεί πραγματικά με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στις διαπραγματεύσεις καμιά φορά η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου δεν είναι πάντα ομόφωνη στην απόφασή της, στη θέση της. Και καμιά φορά υπάρχουν έτσι διαφορετικές τάσεις για το μέχρι πού μπορούμε να πάμε, ποια θα πρέπει να είναι η συμβαστική μας πρόταση. Ο, πρό, πρόεδρος έχει τον ε, ρόλο να βρει ένα κοινό τόπο. Ε, καμιά φορά, κύριε Βαλέσα, υπάρχουν και κάποιοι που δυσαρεστούνται από το αποτέλεσμα. Αλλά τι να κάνουμε, οι συμβιβασμοί έτσι είναι. Στο τέλος όμως και για τους δύο αυτούς φακέλους εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί μπορέσαμε να έχουμε την ρεσιμότητα που θέλαμε, τις ασφαλιστικές δικλείδες που θέλαμε, τις απαιτήσει που είχαμε βάλει για την καλή διακυβέρνηση. Νομίζω ότι ήταν επιτυχία αυτό για το Κοινοβούλιο και για τις ποσοστώσεις. Όντως, ε, έχουμε έναν συμβασμό στο τραπέζι. Αλήθεια είναι αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Βαλέσσα για την σκληρή δουλειά. Ε, κάνατε πραγματικά πολύ καλή δουλειά, εις βάθους ανάλυση, λεπτομερή δουλειά. Τέτοιου είδους δουλειά χρειάζεται το Κοινοβούλιο για να μπορεί να προωθεί την θέση του και να τη μεταφράζει σε πραγματική νομοθεσία. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ο τρίτος τώρα φάκελος είναι το πακέτο εξχρονισμού ε, για, το, για το εμπόριο. Δεν είναι εδώ ο διαπραγματευτής μας. Είχαμε τέσσερις τριμμένες διαλόγους. Και νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να διατηρήσουμε το ορόσημο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας και να προχωρήσουμε και σύντομα να, συνεχίσουμε και με την Εστονική Προεδρία γιατί πήραμε αρκετά, αλλά το πιο αντικρουόμενα ζητήματα για τους διάφορους κανόνες και την άρση των κανόνων για τα περιβαλλοντικά θέματα, για τη ρήτρα, για τις αποστολές, για τους dealers που πρέπει να ενημερώνονται για τους μηχανισμούς, τους αμυντικούς μηχανισμούς. Όλα αυτά δεν καταφέραμε να τα συμφωνήσουμε, δεν έχουμε κάποιο συμβασμό. Οπότε η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί. Και όπως είπα, είμαστε σε πολύ καλή φάση και πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την όθηση που έχουμε και για τα τεχνικά στοιχεία αλλά και για τα πολιτικά. Έχουμε κάποιες προσωρινές συμφωνίες, αλλά βεβαίως τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν συμφωνηθούν τα πάντα. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το φάκελο αυτό και να τον προωθούμε για κατά τη διάρκεια της Εστονικής Προεδρίας. Και μία ανακοίνωση ακόμα. Ξέρατε ότι ο πρώην συνάδελφός μας Ντεσονής είναι ε, Ευρωπαϊκό, είναι υπουργό η κυρία είναι υπουργό ε, Ευρωπαϊκών Θεμάτων στη Νέα Γαλλική Κυβέρνηση. Ε, θα αντικατασταθεί από την κυρία Πατρίσια Αλόντ. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία στα καθήκοντά σα στην Επιτροπή μας. And then we switch to... Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο, σημείο 7, πρόταση για πράξη της Ένωσης σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου στις ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς. Και τα σημεία 8 και 9 επίσης επικεντρώνονται και πάλι στην, στις επενδύσεις, άμεσες επενδύσεις. Και είναι σαφές ότι μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη, το θέμα των αρμοδιοτήτων δεν είναι απολύτως σαφές και δεν έχει κλείσει. Τα κράτη-μέλη πρέπει επίσης να το συζητήσουν. Τώρα για τις δικές μας τις ε, συμφωνίες ε, είναι μεικτή η αρμοδιότητα. Παρ' όλα αυτά η πολιτική για τις ε, επενδύσεις αμυγός αναφέρεται στο άρθρο 207 της συνθήκης. Και είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι. Στο σημείο 7 έχουμε λοιπόν την πρόταση αυτή που αντικατοπτρίζει τις μεγάλες επενδύσεις από συγκεκριμένους εμπορικού εταίρους μας για το προηγούμενο έτος σε στρατηγικού τομεί. Και πρέπει να δούμε πώς θα τη διαχειριστούμε. Η Ολομέλεια στις 14 Ιουνίου την προηγούμενη εβδομάδα συζήτησε το θέμα αυτό και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης θα συζητήσει το θέμα αυτό εντός της εβδομάδος. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που έχουμε τον κανόνα 46.2 και έχουμε μια σχετική πρόταση δυνάμει του κανόνα αυτού στην ε, Επιτροπή μας και θα δώσω το λόγο στον κύριο Πούς, έναν εκ των συγγραφέων της πρότασης, το λόγο για να την παρουσιάσει έτσι όπως την συνέδεξε μαζί με κάποιους συναδέλφους του. Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα εθνικής ασφάλειας αφορά τα κράτη-μέλη σε σχέση με τον πόλεμο και με την τρομοκρατία. Δηλαδή αυτό πρόκειται για την καρδιά δραστηριότητα ενό κράτου μέλου και έχει σχέση και με οικονομία και με και έχουμε ένα τέτοιο δίκτυο επιχειρήσεων και βιομηχανό δίκτυο. Και έτσι κάνουμε τις εξαγωγές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε το know-how και όλα αυτά με κάποιες συνθήκες ασφάλειας, αξιοπιστία και εμπειρογνωμοσύνη, οπότε βέβαια είναι και θέμα επενδύσεων και θα συνεχίσουμε να βοηθούμε τι εξωτερικέ επενδύσει στην Ευρώπη, ακριβώ όπω και εμεί επενδύουμε στο εξωτερικό. Δεν είναι το θέμα του να γλιστρήσουμε σε κάποιο είδου στήρο προστατευτισμό, αλλά είναι θέμα ισορροπία, οπότε και σήμερα ε, με βάση τη λογική μπορούμε να αναρωτηθούμε κατά πόσον έχουμε χάσει την ισορροπία μας μέσω κάποιες απειλής. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Υπάρχει αμοιβαιότητα όσον αφορά τις επενδύσεις για τις επιχειρήσεις μας και υπάρχει επίσης κίνδυνος για την τεχνογνωσία μας όσον αφορά την σχετική μας στρατηγική. Γιατί αν θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις μας έχουν κάποια στρατηγική, τότε θα πρέπει οι εξωτερικές επενδύσεις και αυτές να έχουν στρατηγικό χαρακτήρα. Όταν όμως δεν υπάρχει αμοιβιότητα για τις επενδύσεις, τότε έχουμε μια στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Και αυτό το διαπιστώνουμε πάρα πολύ καλά όσον αφορά την Κίνα. Είδατε τι γίνεται με το China Manufacturing Plan του 15 ε, και αυτό το στήσαμε ακριβώ στο ήταν χαρακτήρας χαρακτήρα γιατί πρόκειται για κάποια χώρα που έχει αυτάρκεια βιομηχανική. Από την άλλη μεριά όμω δεν μπόρεσαμε να έχουμε κάποιο διμερή συμφωνία ε, και χωρί την αμοιβαιότητα αγαπητοί συνάδελφοι Όσον αφορά τι πολιτικέ των επενδύσεων, πώ να θεωρήσουμε ότι οι εμπορικέ συνταλλαγέ διέπονται από δικαιοσύνη. Κάθε μέρα του διαβάζουμε τι εφημερίδε και το βλέπω και στην ε, εκλογική περιφέρεια, το ότι εξαγοράζονται οι επιχειρήσει από κάποια ταμεία. Ε, αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Ε, Προφανώ αυτό μα ανησυχεί και κυρίω διότι έχουμε κάποιε ευαίσθητε τεχνολογίε ή κάποιου ζωτικού τομεί για την ανεξαρτησία, για την ε, ανάπτυξή μα θίγονται. Ε, οπότε θα πρέπει τώρα να μπορούμε να αντιδράσουμε, να σταματήσουμε τον εφησυχασμό. Και οπότε και από το ΕΛΚ προτείναμε να υπάρξει μια πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα. Οπότε αυτό θα πρέπει να προσθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάποια μελέτη για αυτή την κατάσταση και να διατυπώσει προτάσεις, διότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο και ο καθένας ε, να συνειδητοποιήσει ότι αν δεν έχουμε ενία αντίδραση είμαστε όλοι χαμένοι. Γιατί αν ο ένας προστατεύεται πάρα πολύ από τις επενδύσεις, τότε οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσεις σε αυτή τη χώρα θα υποφέρουν γιατί δεν θα υπάρξουν επενδύσεις. Και το αντίθετο, εάν ένα κράτο δεν προστατεύει καθόλου σε με τι επενδύσει, τι ξένε και εχθρικέ τι επιχειρήσει του, ε, τότε δεν θα υπάρξει υπεργολαβία τότε αυτό θα έχει επίσης διακρίσει, ε, επενδύσεις στην Ευρώπη. Είχαμε τρεις υπουργού από Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία και είπαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή ότι θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα. Το θέμα δεν είναι αν θα πρέπει ή όχι να το κάνει η Κομισιόν. Το θέμα είναι πότε θα το κάνει. Πρόκειται για κάποιο πρωτοβουλίο που την ξεκινήσαμε εδώ και στόχο είναι να επιταχυνθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα, όποια και να είναι η σχέση μα, όποιε και να είναι οι απόψει μα. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε αυτή την απόφαση έτσι όπω είναι τώρα σε Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκό επίπεδο να βαδίζει μόνη τη. Θα πρέπει να τοποθετηθούμε, θα πρέπει να ζητήσουμε την Κομισιό να κάνει τι αναγκαίε μελέτε και κυρίω, και σε αυτό επιμένω, να διατυπώσει πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έχουμε τώρα πιο πολλά ερωτηματικά παρά απαντήσει για αυτό το θέμα. Ε, γι' αυτό και είπαμε να λάβουμε αυτή την πρωτοβουλία για αυτέ τι ξένε επενδύσει στα δικού τομεί και τη σχετική πράξη. Και γι' αυτό θέλουμε η Επιτροπή ΙΝΤΑ να επιληφθεί αυτού του σημαντικού ζητήματο που είναι σημαντικό και για τον κόσμο και για τις επιχειρήσεις. Την περασμένη εβδομάδα, ξέρετε, στο Στρασβούργο, θα το θυμάστε πρόεδρες, στην ε, Ολομέλεια, ο Ντανιέλ Κασπαρή ε, είπε με τρόπο που κανείς δεν ξέχασε το ότι είχαμε την διαγύριση του Τζιγκιμπίνγκ, του Κινέζου Πρόεδρου στην αρχή της χρονιάς ότι δηλαδή θα ανοίξει και δεν θα ξανακλείσει ποτέ την πόρτα της η Κίνα. Ε, καλά, ας έχουμε λίγο χιούμορ και θα πρέπει να σας πω ότι δεν μας αρκεί το να μείνουμε στο κατόφλι μόνο. Okay, now Μάλιστα, τώρα λοιπόν θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής, έτσι ώστε να ακούσουμε τις απόψεις τους για την πρόταση αυτή. Τέσσερα μέλη έχουν ζητήσει, πέντε το λόγο, έξι, εφτά, μάλιστα. Οχτώ. και σας παρακαλώ να μην υπερβείτε τα τρία λεπτά. Πρώτη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει κυρία Σάιφη, ναι βεβαίως και συμφωνώ με τα όσα μας ε, είπε ο κύριος προστιθή την ε, πρωτοβουλία. Ε, βέβαια το μήνυμα είναι ξεκάθαρο για την οικονομία μας, αυτές οι ξένες επενδύσεις βοηθούν και στην ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει ε, να παρακολουθήσουμε τα όσα γίνονται και θα σας επιστρέψω την προσοχή σε κάτι πάρα πολύ σχετικό. Μεταξύ 2015 και 2016 οι κινέζικες επενδύσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 77%. Όμως ε, ε, αντιστρόφως οι δικές μας στην ε, η Κίνα συρρυκνώνονται όλο ένα και περισσότερο, άρα θα πρέπει να ξαναβρεθεί η ισορροπία ε, που επιβάλλει η μηβιότητα και θα πρέπει να σταματήσει η Κίνα να πολλαπλασιάζει τους φραγμούς για τις επενδύσεις. Και ο πρόεδρος, όπως είπε ο Φρανκ, είπε ότι ανοίγουν οι πύλες της Κίνας για τους επενδυτές στο τελευταίο Νταβός και περιμένω ε, συγκεκριμένες πράξεις, αλλά προς το παρόν δεν έχω δει τίποτα. Τώρα, όσον αφορά τι επενδύσει στατικού τομεί, υπάρχουν κάποια μέσα και εργαλεία σε κάποια κράτη-μέλη, ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε. Και άρα θα πρέπει ιδίω για θέματα ασφαλείας να μην αναλάβουν τα ενία της άμυνας οι ξένοι ή να μην αναλάβουν τα ενία της ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα πρέσβευε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, σεβασμός, να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμό. Ε, γι' αυτό και θα πρέπει να εναρμονίσουμε την πολιτική μας και να έχουμε ένα μέσο ευρωπαϊκό που να παρεμβαίνει όταν υπάρχει πρόβλημα. Και τέλος για άλλη μια φορά να μην με σταυρωμένα τα χέρια ενώπιον των εξελίξεων. Η αμοιβιότητα θα πρέπει να είναι πυλώνα για την πολιτική επενδύσεων και εμπορική πολιτική. Γενικώ. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που ζητούμε κάτι τέτοιο. Και ελπίζω ότι η πρόταση του ΕΛΚ θα υποστηριχθεί και θα καταλήξει σε πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλό είναι που μιλάμε για τις ε, ξένες επενδύσεις στα πλαίσια του τομέα στρατηγικής της Ένωσης. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να γνωρούμε το πόσο σημαντική είναι η ανάληψη ευθυνών. Είναι καλές οι επενδύσεις, όμως ε, δεν πρέπει να γίνουν δόγμα. Πρέπει να δούμε όλες τις πτυχές τους και πρέπει να καταστήσουμε σαφές ε, το εξή. Φυσικά να πω καταρχά ότι δεν είμαι κατά των ξένων επενδύσεων γιατί προωθούν την ανταλλαγή κεφαλαίου, ιδεών, τεχνολογία κτλ. Αυτό είναι πάντα καλό για την οικονομία. Τα τελευταία χρόνια όμως το επίπεδο επενδύσεων από την Κίνα έχει αυξηθεί και αυτές οι επενδύσεις εστιάζουν σε ένα βαθμό ε, σε σύγχρονες εταιρείες που έχουν πολύ ενδιαφέρουσες ε, τεχνολογίες να πουλήσουν και αυτό φυσικά ε, να μην το πάρουμε και στραβά η Κίνα θέλει να αγοράσει καλές εταιρείες, δεν θέλει να αγοράσει κάτι που δεν είναι καλό και αυτό δεν είναι επιλήψιμο. Όμως η εταιρείε πρέπει να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν σε ποιον θα πουλήσουν και πολλές φορές η τιμή είναι αποφασιστικός παράγοντας. Χρηματοδότηση τώρα. Ένα από τα σημαντικά ε, θέματα που μας προκαλούν ανησυχία με τις ξένες επενδύσεις από την Κίνα είναι ότι πολλές φορές οι αγοραστές ε, είναι δημόσιοι φορείς, είναι από το κράτος. Υπάρχει δηλαδή η αντίληψη, ίσως λανθασμένη, ίσως και όχι, ότι ορισμένες εταιρείε ε, στην Κίνα που αγοράζουν ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία ε, δεν είναι εταιρείε, είναι η κυβέρνηση της Κίνας στην ουσία που αγοράζει μια ευρωπαϊκή επιχείρηση. Μία δηλαδή από τις ε, ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου έχει πρόσβαση σε ε, άπλετη χρηματοδότηση από το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι θα δίνει πολύ καλύτερη προσφορά από οποιοδήποτε άλλον υποψήφιο αγοραστή. Ε, τι θέλω να πω με όλα αυτά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τις ξένες επενδύσεις. Δεν πρέπει φυσικά να ε, είμαστε βιαστικοί, αλλά πρέπει να σκεφτούμε διάφορα και να αναρωτηθούμε τα εξή. Καταρχάς, σε ποιοι τομεί είναι στρατηγική σημασία. Πρέπει να προσέξουμε να μην εμποδίσουμε τις επενδύσεις στην ε, φυσιολογική, αν θέλετε, οικονομία. Μετά, το δεύτερο, ποιος θα διεξάγει τους ελέγχους αυτούς. Διότι με ανησυχεί ε, η περίπτωση να γίνει πάλι αυτό διελκυστήντα δυνάμεων στη, ανάμεσα στις Βρυξέλλες και σε έθνη και σε δυνάμεις. Πιστεύω πως τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν το τι αποτελεί για αυτούς θέμα εθνικής ασφάλειας. Και τώρα, εθνική ασφάλεια. Εθνική ασφάλεια αφορά κυρίως ε, περιορισμένη γεωγραφική επικράτεια. Αφορά ένα κράτος, έχει υπόβαθρο ιστορικό και πολιτικό. Φοβάμαι πως αν δώσουμε υπερβολικά πολλές εξουσίες στις Βρυξέλλες θα ε, ακούσουμε πάλι κατηγορίες ότι οι Βρυξέλλες προσπαθούν να αρπάξουν την εξουσία από τα χέρια μας. Και μετά πρέπει να επιλέξουμε, να επιλέξουμε ε, δικαιοδοσία, γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρξουν και τέτοια θέματα. Μετά, πρέπει να γίνεται μία έρευνα προτού αρχίσει η διαδικασία εξαγοράς μιας επιχείρησης. Έρευνα που να κάνει έναν έλεγχο για θέματα ασφαλείας, για τις πηγές της χρηματοδότησης, αν είναι δημόσια ή ιδιωτική ε, η επένδυση, ποιος θα είναι ο ανάδοχος, όλα αυτά που γύρουν ερωτήσεις. Και τέλος πρέπει να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση των ενδικών μέσων, τι μπορούμε να κάνουμε, εάν θέλουμε να σταματήσουμε μία ε, συναλλαγή, μία εξαγορά, πώς μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται επίσης με τα λόμπι, εάν θα είναι καλύτερο να δράσουμε έτσι ή να προσφύγουμε σε ε, άλλες λύσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά λοιπόν ερωτήματα τα οποία παραμένουν αναπάντητα. Ξέρω πως ο κύριος Προύστ εργάζεται σκληρά και είμαι σίγουρος πως θα ελέγξει την κατάσταση και θα την παρακολουθήσει. Αυτά λοιπόν από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το σχεδόν έλεγα με το κοινό εμπορικό θεματολόγιο. Ε, επιθετικό έχει ο καθένα. Προ τα έξω, αν θα πρέπει να ενισχύσουμε το προστασιό μα. Γι' αυτό αφορά και τι επενδύσει, Γιατί, γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσει την αμοιβαιότητα η Ευρώπη. Το είπαν ήδη οι προλέξατε συνάδελφοι. Οι κινέζικε επενδύσει σε τρία χρόνια τριπλασιάστηκαν και οι δικέ μα. Είναι σε στασιμότητα για να μην μπω σε συρρήγνωση. Επομένω, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τι γίνεται, ποιος, σε ποιο τομέα, σε ποια περιοχή επενδύει. Και αν κάνουν αυτές τις ερωτήσεις, δίνουμε τις απαντήσεις. Όχι. Και για να πετύχουν οι διαπραγματεύσεις με τις τρίτες σχόλες ε, αυτό εξαρτάται και από το πόσο στεγανές είναι οι διατάξεις του ιστορικού μα. Γιατί νομίζετε η Κίνα δεν θέλει να υπογράψει συνεργασία επενδύσεων μαζί μα. Γιατί, γιατί έχουν ήδη πρόσβαση όπου θέλουν απεριόριστη. Γιατί να κάνουν συμφωνία. Επίσης και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν, να καταπολεμήσουν αυτή τον αθέμητο ανταγωνισμό. Άρα να προστατεύσουμε και την απασχόληση και τις επιχείρησεις μας. Ιδάλλως, δεν θα έχουμε δώσει απέναντι σε αυτούς που φοβούνται, στους Ευρωπαίους που φοβούνται. Ε, αυτοί είναι που κατεβαίνουν στο πεζοδρόμιο κατά του ΣΕΤΑ, κατά του ΤΤΙΠ κλπ. Εμείς, αυτή είναι η δουλειά μας, να προστατεύσουμε αυτά τους τα θεμελιώδη συμφέροντα. Σαφώς τα έχει προτείνει η πολιτική μας ομάδα νομοθετική πρόταση, ανακλάδο, αμοιβιότητα, έλεγχος. Αλλά αμερικάνικα. Αυτό πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πρόεδρε να σας πω ότι για άλλη μια φορά στην Επιτροπή μας ευτυχώς μπορούμε να συζητήσουμε το πόσο χρειάζεται να έχουμε κανόνες του παιχνιδιού που να είναι ισορροπημένοι. Εδώ και πολύ καιρό το λέμε όλες οι πολιτικές ομάδες. Χρειάζεται αμοιβαιότητα σε αυτούς τους κανόνες του παιχνιδιού για το, για το εξωτερικό εμπόριο. Πάντοτε ήθελε να έχει αντικό πνεύμα, να είναι δίκαιη η Ευρωπαϊκή Ένωση και διμερός και πολυμερός. Αλλά θεωρούμε ότι χρειάζεται η συζήτηση να καταλήξει σε συγκεκριμένα μέτρα που να οδηγήσουν τέλος πάντων σε διαφορετικά μέτρα από αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα δεν έχουμε ισορροπή αντιμετώπιση. Όπω είναι η κατάσταση, μα οδηγεί σε κάποια πόλωση στη διεθνή σκηνή. Από τη μια μεριά έχουμε τη ΣΥΠΑ, που απεμπολεί τι ευθύνε τη στο διεθνέ εμπόριο, στη διεθνή σκηνή. Δεν θέλει δίκαιε ρυθμίσει. Την άλλη μεριά έχουμε την Κίνα Μπράβο που άλλαξαν ε, στάση, μπράβο για αυτά που είπανε, που θέλουν ε, ανοιχτή στάση, πολυμερείς ε, σχέσεις και μακάρι τα λόγια τους να γίνουν και έργα. Να δούμε. Τι θα κάνει η Κίνα, θα τηρήσει τους κανόνες του ΠΟΕ. Θα δεσμευτεί οριστικά. Θα πρέπει να καταλάβουν οι εταίροι μας ότι ήρθε η ώρα να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα. Δεν ωφελούν πια τα ωραία λόγια. Θα πρέπει να περιοριστούμε το μοντέλο μας με αντίστοιχους κανόνες, δίκαιους. Χρειάζεται αμοιβαιότητα όσον αφορά την προστασία του ανοίγματο της πολυμερής σχέσης και όσον αφορά επίσης τις ε, δημόσιες συμβάσεις. Κάθε μέρα τα βλέπουμε αυτά το πόσο χρειάζονται. Βλέπουμε τι κάνουν οι εταίροι μας που δεν συμμερίζονται τις ίδιες ε, αρχές, ούτε δουλεύουν με τους ίδιους κανόνες. Τις προάλλες, ή τέλος των πρώτων λίγους μήνες, με την ευκαιρία να κάνουμε κάποια ανταλλαγή απόψεων και πάλι με τον πρόεδρο του εμπορικού επιμελητηρίου της κοινωνικής και μας είπε ότι συνεχίζουν και υπάρχουν δυσκολίες, τα είπε και η πρόεδρος ότι υπάρχει θέμα με αυτές τις επενδύσεις. Αυξάνονται οι κινέζικες εδώ και μειώνονται οι δικές μας στην Κίνα. Άρα δύσκολα. Επομένω, χρειάζονται κάποια μέτρα που να παρασχούν εγγύησεις για τις στρατηγικές επενδύσεις και με εγγύησει που σημαίνουν ότι δεν θα κινδυνεύει ούτε η βιομηχανία μας, ούτε οι εργαζόμενοι δικοί μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σάκη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να πω πως είμαι ελαφρώς ε, μπερδεμένη. Δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα της συζήτησης. Άκουσα τους συναδέλφους και είχα την εντύπωση ότι το θέμα είναι οι ξανές επενδύσεις σε δικούς μας στρατηγικούς τομείς, όχι διαφορετικό θέμα. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε σαφείς. Τώρα, Προφανώς και πιστεύω πως πρέπει να υπάρχουν κανόνες που διέπουν το εμπόριο και τις ε, επενδύσεις. Γνωρίζω πως υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι στο παρελθόν δεν συμφωνούσαν με την ύπαρξη κανόνων και τώρα ξανασκέφτονται την άποψή τους. Είναι πολύ σημαντικό να μην ε, δράσουμε βιαστικά αλλά να μην είμαστε και αφελείς. Δεν θα έπρεπε να ε, συζητήσουμε τον όγκο των επενδύσεων ή την αμοιβαιότητα όσο το πώς θα διασφαλίσουμε ξεκάθαρα ε, κριτήρια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποιοι τομείς θεωρούνται στρατηγικοί, νευραλγικοί, αλλά όχι μόνο για μας και για τους ε, εταίρους μας και τους συμμάχους μας. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε ε, εκεί. Τώρα, επενδύσεις σε στρατιωτικό τομέα, σε αντικείμενα διπλής χρήσης. Αυτά ήταν πάντα τομείς ευαίσθητοι που και θα έπρεπε να διεξάγονται οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν. Ε, δεδομένης της εξέλιξη της τεχνολογίας ε, και, της ε, μη ευδιάκριτης, και του μη ευδιάκριτου διαχωρισμού ανάμεσα στη στρατιωτική και την πολιτική χρήση νομίζω πω είναι πολύ σωστό να είμαστε επιφυλακτικοί. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο κόσμο αλλάζει ταχύτατα και μαζί με αυτόν και οι τομεί που θεωρούνται στρατηγική σημασία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κάποιες προτάσεις που θα αφορούν τον προστατευτισμό ή κάποια ανάλογα μέτρα. Αλλά ας μην συγχέουμε αυτά τα μέτρα με το γενικό μας ε, στόχο. Ελπίζω, ε, πιστεύω επίσης ότι θα μας βοηθήσουν ε, και διάφορα case studies που θα μελετήσουμε κατά περίπτωση τι έχει συμβεί. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην κάψουμε τα χλωρά μαζί με τα ξερά και να γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννικ. Ευχαριστώ. μία φορά έχουμε, μία μεριά με το TDI, το MS και διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά ότι είναι κάπως αφελής η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αναγκαία συνέπεια, συνεκτικότητα πρέπει να έχουμε και εγώ από πλευρά των πρασίνων. Καταψήφισα την πρόταση Μπαρνιέ για την αμοιβιότητα όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Όχι γιατί δεν πιστεύω στην αμοιβιότητα, αλλά η ιδέα ήταν το να υπάρχει μια αμοιβιότητα και ταυτόχρονα να εγκαταλειφθεί κάποιο μέσο ε, χρήσης και εκμετάλλευσης των δημοσίων αγορών για στρατηγικούς τομείς. Επομένω, αυτό είναι το θέμα. Θα πρέπει με την αμοιβιότητα στις δημόσιες αγορές να κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικός τομέας Έχουμε κοινή εμπορική πολιτική, δεν έχουμε κοινή εμπορική διπλωματία και έχουμε εγκαταλείψει τη φωτοβολταϊκή μας βιομηχανία γιατί υπήρχαν αποκλίνοντα συμφέροντα εθνικά και οπότε είχαμε ε, εκατοντάδες ε, θέσεων απασχόλησης που έτσι διακυβεύθηκαν. Από την άλλη μεριά χαιρόμαστε να έρχεται εδώ μια κρατική κινέζικη εταιρεία και να ασχολείται με ε, την κλοπή πολλών ιδεών εμπορικών. Είδατε τι έγινε και με την EDF. Και εκεί η κυβέρνηση χάρηκε για τις κινέζικες επενδύσεις. Δεν τους αρκούσαν οι ευρωπαϊκές. Οπότε για άλλη μια φορά εμείς συζητάμε για τις επενδύσεις και την Κίνα και κάποιες πολιτικές ομάδες, ακόμα και εκείνοι που σήμερα ζητούν περισσότερο ευφύ αντιμετώπιση της ε, στρατηγικής για τις ξένες επενδύσεις και ζητάτε και δικαστήρια και διατησία και να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ επενδυτών και κράτους. Ναι, σύμφωνοι. σε σχέση με την πρόταση του ΕΠΕ για να υπάρχει πραγματική λογική και συνεκτικότητα όσον αφορά αυτές τις επενδύσεις και αυτό δεν αφορά μόνο την Κίνα. Το Πρόβλημα με την Κίνα έχουμε γιατί το κράτος έχει όπως και το Κατάρ και άλλες χώρες πλεόνασμα ε, δισεκατομμυρίων και ε, οπότε όλα ε, αυτά τα, τα χρήματα έρχονται εδώ μεταμφιεσμένα σε επενδύσεις. Χέλμουν Σόλτς, ευχαριστώ. Συμφωνώ. Είναι ενδιαφέρον ότι στο σημείο 3 το ΕΛΚ έχει ανακαλύψει το δημόσιο τομέα για να επιβάλλει διατάξεις προστασίας. Ε, νομίζω ότι ε, δεκαετίες ή τέλος πάντων χρόνια το ζητά αυτό η αριστερά στην Ευρώπη. Ίσως να είναι λίγο ατυχής η διατύπωση, αλλά νομίζω ότι ε, θα πρέπει να σκεφτούμε τα θέματα αυτά. Ίσως να πρέπει να αλλάξουμε λίγο το πώς έχει η πρόταση. Γιατί δηλαδή να μην επενδύσει κανεί στην ε, δική μα την οικονομία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία, από εταιρείε, από τον δημόσιο τομέα, από κράτη. Μιλάμε για την πολιτική λιτότητα και απ' την άλλη ε, ε, είμαστε έκπληκτοι που δεν έχουμε χρήματα για, την, για τις υποδομές και δεν μπορούμε να κάνουμε τους απαραίτητους εξοπλισμούς. Γιατί να μην τα καταφέρουμε λοιπόν. Γιατί με, το πρόεδρο, με, τον, ε, με το σχέδιο Juncker δεν ε, καλούμε τους Κινέζους να τους πούμε είμαστε μια ανοιχτή αγορά, επενδύστε, εφόσον εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε τα δικά μας λεφτά. Είναι ένα ερώτημα αυτό, γιατί ε, τελικά δεν ξέρει η δεξιά τι πει η αριστερά. Πρέπει λοιπόν αυτή την πρόταση να τη χρησιμοποιήσουμε και εξετάζοντας ακριβώς αυτή την πρόταση να ξανασκεφτούμε η βιομηχανική πολιτική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς θα προχωρήσει, πώς θα, δούμε, πώς θα προχωρήσουμε με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πώς θα επενδύσουμε στις επιστήμες, έτσι ώστε να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο, χρόνο, ε, μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μίλησα για τα διπλώματα. Το 2000, όχι, το 85 η Ιαπωνία ήταν μια χώρα που είχε 257 περίπου χιλιάδες ε, ε, διπλώματα. Η Κίνα είχε 4.000 περίπου, η ε, Γερμανία 45.000, η ΙΠΑ 46.000. Η Γερμανία ήταν τρίτη, στην τρίτη θέση, η Κίνα αρκετά πιο κάτω. Το 2015 στην Κίνα ή δηλώσεις διπλωμάτων για συγκεκριμένους ε, ευαίσθητους τομείς και επενδύσεις έχουν ένα εκατομμύριο και πάνω. Η ΕΠΑ 529, 623. Ε, Η Ιαπωνία 55.000. Νότια Κορέα 288.000. Γερμανία 500.000. Ε, από πρώτο κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την γενοτομία ας πούμε. Θέλω δηλαδή να καταστήσω σαφές ότι οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε πώς προχωρούμε με τη βιομηχανία και με τη μελλοντική ε, πολιτική, αν θέλουμε να μιλούμε για ε, καινοτόμα πολιτική. Και επίσης, τα συνδικάτα οι επενδύσει της Κίνας, ε, είτε είναι της Ιαπωνίας, είτε είναι των ΗΠΑ, στην οικονομία, είναι οι πιο σταθερές ό,τι αφορά την δημιουργία θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ, θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα. Κυρίως γιατί θα πρέπει κάπως να διαχειριστούμε αυτές τις επενδύσεις που είναι λόγια και πιο σημαντικές. Και σήμερα Επομένως, βλέπουμε ότι είναι ακόμη πιο καυτό το θέμα. Μια που έχουμε επενδύσει από χώρες που δεν έχουν την ίδια δημοκρατικότητα και διαφάνεια. Α, η Κίνα. «35 δις, 77% ασχέσεις με πέρσι αυξήθηκαν οι κινέζικες επενδύσεις. Βέβαια βοηθούνται έτσι σε δύσκολες ώρες. Η, αυτό ήταν επνοή ζωή για τι επιχείρησεις μα. Όμως, τι θα γίνει μετά. Η Κίνα δεν είναι οικονομία τη αγορά. Είναι κεντροκατευθυνόμενη οικονομία. Όλα κινούνται από το Πεκίνο. Να δούμε τι θα γίνει με όλα αυτά τα στρατηγικά ατού, τις στρατηγικούς τομείς. Ας πούμε τι γίνεται με την τεχνολογία εχμής. Δεν θα πρέπει να φεύγουν από την Ευρώπη αυτές οι βιομηχανίες είναι επομένω το θέμα πιο πολύ πολιτικό παρά οικονομικό. Ειλικρινά σας λέω, αυτές οι επενδύσεις είναι αρμοδιότητα τη Ένωσης. Επιβάλλεται έλεγχος. Να δούμε τι γίνεται με τις δεσπόζουσα θέση, με τον ανταγωνισμό, όλα αυτά. Να τα εξετάσουμε. Τι γίνεται πλευρά ασφάλειας. Αλλά το κάθε κράτος μέλος δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά. Ακόμα και όταν έχουμε και κρατικές ενισχύσεις. Είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας, προστασία του περιβάλλοντος, αλλά όμως πολλές φορές αυτές οι ενστάσεις δεν πιάνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης. Γιατί πάντοτε λέμε ότι κατησχεί η ελευθερία των επενδύσεων. Τι μπορούμε να κάνουμε μπορούμε ε, να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη και έτσι να πάνε σε πιο προστατευτικές θέσεις. Ίσως αυτό θα μπορούσε να γίνει με το σημερινό νομικό πλαίσιο. Αν όχι, έας τροποποιηθούν οι συνθήκες. Άλλη λύση. Να έχουμε ένα κοινοτικό μέσο έλεγχες, μια επιτροπή ειδικών και περιπτωσιολογικά να κρίνουν α, την κάθε τέτοια επένδυση. Όπως της είπα. Αλλά να δούμε ότι έτσι θα πρέπει να αξιολογήσουμε το να... Δεν πρέπει έτσι να έχουμε ε, κάποιες ε, στρατηγικές ξένες επενδύσεις. Να μην κατησχύει επομένως χωρίς προβληματισμό πάντα η ελευθερία της επένδυσης. Πολλές φορές οι επενδύσεις δεν έχουν μόνο οικονομικό σκοπό. Να υπάρχουν επίσης εγγυήσεις αντιπροσωπευτικότητας. Ποιοι θα συμμετάρχουν σε αυτές τις επενδύσεις, μόνο ξένοι ή και Ευρωπαίοι. Και εδώ είναι θέμα δημοσίου συμφέροντος αυτή η αντιπροσωπευτικότητα, η συμμετοχή. Και βέβαια αμοιβαιότητα σημαίνει το όλα αυτά που λέμε που ισχύουν για τους ξένους επενδυτές να τα εφαρμόσουν και ξένοι για τις δικές μας επενδύσεις στη χώρα τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάρχη μου Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριο Σούστερ. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή τη συζήτηση. Είναι απόλυτα δικαιολογημένα τα επιχείρηματά σα. Ωστόσο, ελπίζω να μην μείνουμε στα μέσα του δρόμου, να φτάσουμε μέχρι το τέλο. Χρειάζεται να καθορίσουμε τα στρατηγικά μα ενδιαφέροντα, διότι αυτή τη στιγμή η παγκόσμια οικονομία χαρακτηρίζεται από διάφορε δυνάμει που μα τραβάνε. Η Ασία αυτή τη στιγμή ανεβαίνει πάρα πολύ και η εθνική οικονομία στην Κίνα ακολουθεί ένα τελείω διαφορετικό μοντέλο εξέλιξη από ότι εμεί. Οι εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της Κίνας λοιπόν ελέγχονται πάρα πολύ, διέπονται από αυστηρού κανόνες, ελέγχονται από το κράτος. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλο επίτευγμα το ότι μας δέχονται στη χώρα τους. Και ε, είναι απόλυτα λοιπόν κατανοητό το ότι στηρίζουν πάρα πολύ τις ε, δικές τους επιχειρήσεις. Ε, νομίζω πως πρέπει να δούμε εάν υπάρχουν θέματα ε, εθνικής ε, ασφάλειας, εάν υπάρχουν επενδύσεις που αφορούν τους τομείς ασφάλειας και να δούμε τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Ε, στο τέλος πρέπει να διερωτηθούμε ποια είναι η βιομηχανική πολιτική που ακολουθούμε και τι θέλουμε. Η βιομηχανική πολιτική τα τελευταία χρόνια ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Στην ουσία ακολουθούσαμε το δόγμα της ελεύθερης αγοράς, το οποίο δόγμα όμως ε, αποδεικνύεται όλο ένα και ε, λιγότερο αποτελεσματικό, διότι βλέπουμε στην Ασία να αναδύονται νέα μοντέλα, τα οποία είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι σε αυτή τη ε, δημόσια συζήτηση δεν πρέπει να μείνουμε στο, στα στενά πλαίσια της εθνικής ασφάλειας, αλλά να δούμε ποια είναι τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν κόσμο που αλλάζει ε, με ταχύτητα τους ρυθμούς. Ποιοι είναι οι τομεί που πρέπει να προστατευτούν από εμάς, ποιοι είναι οι τομεί που πρέπει και μπορούμε να αναπτύξουμε και πώς θα διαμορφωθεί η σχέση μας με την Κίνα ε, ως εκ τούτου. Νομίζω ε, δεν πρέπει να μιλάμε για προστατευτισμό, αλλά πρέπει να εντοπίσουμε τους ε, νευραλγικούς τομείς ε, στρατηγικά μιλώντας και να δούμε τι είναι επίκαιρο. Αυτή τη στιγμή ο χάλιβα, η βιομηχανία χάλιβα είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Υπάρχουν προστατευτικά μέτρα τα οποία έχουμε υιοθετήσει για ε, την προστασία του, ε, της βιομηχανίας μας. Για, ε, μιλάμε για κάποιες χιλιάδες θέσεις εργασίας, όμως η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε και η συμπεριφορά μας θα επηρεάσει και άλλους τομείς. Δεν ε, είναι μόνο κάτι που αφορά στενά κάποια συνδικάτα, κάποιου συνδικαλιστέ σε μία μικρή μερίδα τη βιομηχανία μα. Είναι λοιπόν θέμα και βιομηχανική πολιτική. Πρέπει να το συζητήσουμε και να βρούμε στο τέλο και μία απάντηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τελευταίο έχει το λόγο η κυρία Όχι. Ο κύριος Σάινφελντ. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Πρόεδρε, αυτό το θέμα ίσως δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είναι περίπλοκο. Και τη σήμερα ημέρα τα οικονομικά συμφέροντα και τα συμφέροντα των κρατών αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοσυσχετίζονται. Δυστυχώ, μερικές χώρες εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις και τα πράγματα χειροτερεύουν. Άλλες χώρες έρχονται κάποιες πρακτικές επομένως που δεν είναι σωστές, ε, οπότε γι' αυτό και αυτή η πρόταση για πράξη της Ένωσης σχετικά με το θέμα είναι πάρα πολύ σωστό. Θα πρέπει όμως πριν εγκρίνουμε μια τέτοια πράξη να καθορίσουμε με ποια κριτήρια κάποια επένδυση συνάδει με την αρχή της ελεύθερης αγοράς, με την ασφάλεια που θέλουμε να έχουμε, γιατί έχει πολλές όψεις η ελεύθερη αγορά. Θα πρέπει επομένω να ορίσουμε κάποια κριτήρια. Βάσει αυτό να κρίνουμε εάν κάποια επένδυση έρχεται σε αντίθεση με τις δημοκρατικές αρχές μας για την οικονομία. Ακόμα και σε περιπτώσει που θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνε ή ίσω δεν παραβιάζονται οι δημοκρατικέ αρχέ και ενώ σε άλλε περιπτώσει το αντίθετο. Επομένω, το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή θα πρέπει να κρυθεί το τι σκοπούς έχει κάθε χώρα με τις επενδύσεις της. Είναι επικίνδυνη αυτή η σκοπή ή δεν είναι αλλά θα πρέπει να κρίνεται κάθε φορά ο σκοπός της επένδυσης. Βέβαια ο καθένας έχει άλλους, άλλες μεθόδους, άλλους τρόπους να εισδύσει σε κάποια αγορά. Δεν το ξέρουμε αυτό με τους εταίρους μας. Ο, η Γαλλία ας πούμε πολλές φορές ε, έχει εταίρο κάποια άλλη εταιρεία και δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές κάποιος προσπαθεί να διεισδύσει μέσω ε, ε, κοινοτικής εταιρείας, όχι εξωκοινοτικής. Είναι πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς το τι γίνεται. Επίση, επίσης, έχουμε και ίδρυση εταιριών από κάποια τρίτη χώρα, αλλά η έδρα της είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται αυτό στο Λουξεμβούργο, στην Ελβετία και αυτές οι εταιρείες ασχολούνται με ευαίσθητους τομείς, τους στρατηγικούς τομείς. Άρα, προσοχή, προσοχή. Γιατί βλέπω να δεκρίνει τη συζήτησή μας υπερβολική αισιοδοξία. Προσοχή. Deputy Head of Unit. Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Κάρλο Πετινάτο από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα απαντήσω σε κάποια από τα σχόλια που έκανε ο Επίτροπος Μοσχοβησή την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Εμείς ακούμε αυτά που λένε τα κρατημέλη, αυτά που έχουν προτείνει. Ακούμε τι λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποιες είναι οι απόψεις σας. Είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα και υπάρχουν αρκετές ανησυχίες, όχι μόνο μία, αρκετές. που δημιουργούν την ανάγκη να, ελέγχει, να υπάρχει μια, ένας έλεγχος για τις ε, ξένες επενδύσεις. Είναι περίπλοκο λοιπόν το θέμα. Αναλύουμε εντός των παραμέτρων του υπάρχοντος νομικού πλαισίου που έχουμε τα πράγματα, όχι μόνο δηλαδή τη συνθήκη, δεν εφαρμόζουμε ε, πολιτική εμπορική στο κενό, έχουμε διάφορες ε, διεθνείς υποχρεώσεις που μας δεσμεύουν, οπότε εντός αυτού του πλαισίου προσπαθούμε να δούμε ποια εργαλεία έχουμε και πώς μπορούμε να απαντήσουμε στις ανησυχίες. Κάποια σχόλια. Το θέμα της αμοιβαιότητας βεβαίως ε, προκύπτει συχνά, υπάρχει και στην πρόταση να υπάρχει μια πράξη της Ένωσης σχετικά για να επιτύχουμε έτσι μια ισότητα όπλων με τους εταίρους μας. Είναι στον πυρήνα της πολιτικής εμπορίου βεβαίω αυτό και κυρίως ό,τι αφορά την Κίνα και τις διαπραγματεύσεις που κάνουμε. Ε, η προσπάθεια αυτή είναι συνεχής. Οι διαπραγματεύσει δεν έχουν τελειώσει και η βασική εντολή που μας έχουν δώσει τα μελη είναι ακριβώ να επιτύχουμε καλύτερη πρόσβαση στην αγορά και να προσπαθήσουμε να έχουμε ε, ένα, μια ισοτιμία ε, όπλων. Επίσης, να δούμε και τις υπόλοιπε χώρε Το αμερικανικό μοντέλο, που πούμε, αναφέρθηκε αρκετά. Θέλω να σημειώσω ότι το αμερικανικό μοντέλο δεν περιλαμβάνει και κανένα άλλο μοντέλο, δεν περιλαμβάνει το κριτήριο της αμοιβαιότητας ως κριτήριο ε, για την σύναψη των συμφωνιών και τις ξένες επενδύσεις. Οπότε αυτό το έχουμε υπόψη. Επίσης, ε, διαπραγματευόμαστε την ε, συμφωνία αυτή με την Κίνα που θα επιτρέψει στους Κινέζους επενδυτές να χρησιμοποιούν ιδιωτικά δικαστήρια. 27 ε, κρατημέλη υπάρχουν που έχουν διμερείς συμφωνίες με την Κίνα που ήδη σήμερα δίνουν πρόσβαση στους Κινέζους, στους Κινέζους επενδυτές για την, στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών κρατών και επενδυτών. Οπότε από εκεί πορεύει και η πρόταση για το νέο σύστημα αυτό του Διεθνούς Δικαστηρίου Επενδύσεων. Ε, μελετούμε λοιπόν ε, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα δούμε αν θα υπάρξει πολιτική απόφαση για να γίνει κάτι. Αν υπάρξει βεβαίω θα παρουσιάσουμε και εμεί σχετικά τι ιδέε μα. Ευχαριστώ. Οι συντονιστέ θα συζητήσουν σήμερα τη διαδικασία και πώ θα διαχειριστούμε την πρόταση αυτή. Νομίζω θα έχουμε πολλές συζητήσεις ακόμη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ όλους. Πάμε στο σημείο 8. Μιλήσατε για το ISDS, το σύστημα ε, επίλυσης διαφορών κρατών επενδυτών. Το ε, Κοινοβούλιο αποφάσισε να αφαιρέσει το σημείο αυτό από όλες τις εμπορικές συμφωνίες και θα ζητήσουμε ένα νέο σύστημα για την επίλυση διαφορών μεταξύ δημοσίου τομέα και επενδυτών. Οι που πριν από κάποιους μήνες αποφάσισαν να, κάνουν, να γίνει μια μελέτη για αυτό το νέο μέσο, το νέο εργαλείο. Ζητήσαμε από έναν εμπειρογνώμονα περί επενδύσεων που έχει δουλέψει αρκετά με το Κοινοβούλιο και τα θέματα επενδύσεων να εκπονήσει αυτή τη μελέτη και είναι τώρα εδώ μαζί μας για να μας παρουσιάσει αυτό το σχέδιο έκθεσης για την ε, δημιουργία ενός ε, ε, διεθνούς δικαστηρίου επενδύσεων. Είναι ο καθηγητής Χίντενλανγκ από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να μου να παρουσιάσω ότι τα βασικά ευρήματα αυτής της έκθεσης, να κάνω κάποια, θα κάνω και βέβαια κάποια σχόλια για την απόφαση του δικαστηρίου για την Σιγαπούρη. Η μελέτη συγκρίνει τη ΣΕΤΑ, το, την ε, Συμφωνία Ελεύθερου με το, με το Βιετνάμ και την ε, Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τη Σιγκαπούρη σε ό,τι φορά την ε, δυνατότητα και τις διατάξεις που υπάρχουν για την επίλυση διαφορών με τους επενδυτές. Υπάρχει βεβαίως αντιπαράθεση με τους διαδικαστικούς κανόνες που εφαρμόζονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. η μελέτη προσπαθεί να δώσει ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της ε, πρόοδου που έχει γίνει ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση του καθεστώτος του Διεθνούς Δικαίου για τις Επενδύσεις και επίσης δίνει στα μέλη του Κοινοβουλίου και στο ευρύ κοινό βέβαια ένα εγχειρίδιο για να κατανοήσουν την, και να αξιολογήσουν την μελλοντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες. Έχουμε κάποια βασικά στοιχεία της ε, διαδικασίας που έχουν να κάνουν με, με δύο υπάρχοντα συστήματα και επιτυχώς λειτουργούν τα δικαστήρια ουσιαστικά. Από εκεί πήραμε την έμπνευσή μας για το νέο αυτό ε, δικαστήριο. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σε διαφορά την πρόοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού καθεστώτος για, το, ε, για την νομοθεσία για τις επενδύσεις. Έχουμε την ε, παραδοσιακή προσέγγιση για την ε, διαμεσολάβηση, για την επίλυση διαφορών επενδυτή κράτους. Είναι μάλλον εξελικτικά και όχι επαναστατικά όσα προβλέπονται εκεί. Και βεβαίως όλες οι ε, συμφορίες ελεύθερου εμπορίου έχουν την πιο παραδοσιακή προσέγγιση από την δεκαετία του 50 και μετά επαφίεται σε κάποιο είδους διαμεσολάβηση για την επίλυση των διαφορών μεταξύ κράτους και επενδυτού. Αλλά αυτή η προσέγγιση παραδοσιακή τροποποιείται κατά τη και συμπληρώνεται από κάποια καινοτόμα στοιχεία, από, την, από, ευρωπαϊκά, από ευρωπαϊκούς κριτές, και, ευρωπαϊκά, ε, και άλλα ευρωπαϊ... Ε, δικαστήρια ευρωπαϊκών χωρών. Προσπαθούμε βεβαίω να απαντήσουμε και στα διάφορα επικριτικά σχόλια για τη διαμεσολάβηση. Προσπαθούμε να καλύψουμε διάφορα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα που θέλουν να διατηρήσουν το παλιό καθεστώς και να καλύψουμε κάποια κενά που υπάρχουν για τι πρακτικέ διαμεσολάβηση σε ό,τι αφορά ε, το κράτο δικαίου. Γενικώ, το τρέχον κείμενο τη Συμφωνία με τη Σιγκαπούρη δείχνει ε, περισσότερα στοιχεία της παραδοσιακής προσέγγισης που βεβαίως έχουν να κάνουν με την ορίμανση των ε, διατάξεων της, των συνθηκών που υπάρχουν. Η ΣΕΤΑ και η Συμφωνία με το Βιετνάμ είναι πιο ουσιαστικές ε, μεταρρυθμίσεις. Πολλά, ε, πολλές από τις καινοτομίε που υπάρχουν στην πρόταση της Κομισιόν για το Διατλαντικό Εμπόριο και τη Σχετική Συμφωνία έχουν ε, ε, παρισπρίσει και στην ΣΕΤΑ και στη συμφωνία με το Βιετνάμ. Επίσης η ΣΕΤΑ και, η συμφωνία με το Βιετνάμ δεν έχουν μόνιμα δικαστήρια για την ε, επίλυση διαφορών. Το νέο ρυθμιστικό καθεστώς για τη ΣΕΤΑ και το Βιετνάμ δεν καλύπτει τη φιλόδοξη διάταξη που προτείνει στην πρόταση της η Κομισιόν για τα αποτελέσματα της συμφωνία. Αλλά η μεταρρύθμιση μάλλον το ποτήρι της μεταρρύθμισης είναι μάλλον μισογεμάτο παρά μισοάδιο. Όλα τα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορές δεσμεύονται από το παλαιό σύστημα επίλυση διαφορών μέσω της διαμεσολάβηση. Όλες οι συμφωνίες ελεύθερης, ε, ελεύθερου εμπορίου συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ad hoc δικαστήρια και παραμένουν ε, συντηρητικοί σε διαφορά τη χρήση εσωτερικών κρατικών δικαστήριων. Ε, επίσης ε, υπάρχουν κάποιοι ε, κριτές, διαιτητές που επιλέγονται από τα κράτη. Προσπαθούμε να αυξήσουμε την διαφάνεια, να είναι τυχαία κατανομή των υποθέσεων, να υπάρχει δημόσια πρόσβαση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μεταρρυθμίσουμε το παλαιό καθεστώς. Το, η τρέχουσα κατάσταση μάλλον δεν θα οδηγήσει, δεν θα είναι η τελευταία σε ό,τι αφορά τι μεταρρυθμίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάποιου μεσοπρόθεσμου στόχου ε, και κάποια βήματα πρέπει να γίνουν για τη δημιουργία αυτού του συστήματο. Η δημιουργία ενός μόνιμου πολυμερούς ε, δικαστηρίου επενδύσεων θα είναι μάλλον ένας μεσοπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος στόχος. Άλλα θέματα που μπορούν να λυθούν ε, πιο άμεσα είναι η συγκεκριμένη κατάσταση που επικρατήσει ότι φορά τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο, στο διεθνές εμπόριο και στι επενδύσεις. Οι, οι συμφωνίες αυτές είναι, μάλλον δεν βλέπουν την πραγματική κατάσταση και την ανομοιογένεια που υπάρχει στους όρους μπορεί κυρίω κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην ε, επωφελούνται από αυτόν τον ε, μηχανισμό διαφορών σε αυτή τη ε, συμφωνία ελεύθερου με τον ίδιο τρόπο που επωφελούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει μια κίνηση προς, μια, προς ύπαρξη κριτών, διαιτητών μόνιμων και με συγκεκριμένη θητεία έτσι ώστε να αποφεύγονται σύγκρουση συμφερόντων. και έτσι δεν θα υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σοβαρή σε ό,τι αφορά την επίλυση διαφορών όταν ε, προσπαθεί να εξασκήσει ε, δημόσια εξουσία στην Ευρώπη. Εδώ το Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει τα ενία και να δημιουργήσει ένα, μια διαδικασία επιλογής για τους μελλοντικού δικαστές. Μόλις λοιπόν γίνει αυτή η διαδικασία μπορούμε να ε, αποκαταστήσουμε την ε, εμπιστοσύνη στους ε, δικαστές και μπορούμε να στείλουμε ένα σωστό μήνυμα, δυνατό μήνυμα, ότι η επιλογή των δικαστών ανεξάρτητα από το που βρίσκονται στο δικαστήριο, είτε στο δικαστήριο ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων, είτε σε οποιοδήποτε άλλο φορέα επίλυση διαφορών, θα πρέπει να είναι το, ε, θα να είναι το ε, δικαίωμα του Κοινοβουλίου να το πράξει. Και επίσης οι συμφωνίε αυτές θα πρέπει να ξανασκεφτούν τη σχέση που έχουν με τα δικαστήρια των κρατών μελών. Η επίλυση διαφορών δεν είναι μονόδρομος, ούτε ο μηχανισμός αυτός είναι μονόδρομος. Αυτός ο μηχανισμός επίλυση διαφορών έχει να κάνει, ε, μάλλον πρέπει να μετατραπεί σε ένα ε, ολιστικό σύστημα επίλυση διαφορών και πρέπει να είναι ε, συγκρίσιμο με, τα, με τους μηχανισμούς που υπάρχουν σε επιμέρους κράτη-μέλη προσπαθώντας να υπάρξει μια ισορροπία για, τα, για το δημόσιο συμφέρον αλλά και το ιδιωτικό. Γι' αυτό είναι πλέον ώρα να επικεντρωθούμε στις σχέσεις της ε, διαμεσολάβησης ε, και των ε, δικαστηρίων στα κράτη-μέλη. Και επίσης, αν επιτρέψουμε έναν τέτοιο μηχανισμό, θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν δικαστήρια που έχουν κερδίσει το σεβασμό των κρατών μελών για την απόδοση δικαιοσύνης σε όλα τα χρόνια που λειτουργούν. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να αποκλείσουμε αυτά τα δικαστήρια από την ε, απόδοση δικαιοσύνη σε τέτοιε περιπτώσει. Μόνο σε διαφορετικέ περιπτώσει μπορεί να έχει ένας επενδυτή πρόσβαση σε αυτά τα δικαστήρια. Σε αυτή την περίπτωση οι Ευρωπαϊκές Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ε, διακήρυξη των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετά υπάρχει και ένας άλλος λόγος γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να σκεφτεί την προσχώρηση σε αυτές τις τοπικές λύσεις. Υπάρχει το προηγούμενο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συγκαπούρης. Υπάρχει γνωμοδότηση σχετικά και αυτή είναι αρκετά διφορούμενοι. Το δικαστήριο λοιπόν υποφάνθηκε ότι ο μηχανισμός διαιτησίας όπως αυτό στην περίπτωση Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Σιγκαπούρης που αφήνει στον επενδυτή να επιλέξει ανάμεσα στα εγχώρια ένδικα μέσα ή στη θεσμική ιδιαιτησία, χρειάζεται τη συγκατάθεση του κράτους μέλους. Επομένως, το καθεστώς ε, που αφαιρεί αυτήν ε, την ε, δυνατότητα από τις δικαιοδοσίες των κρατών μελών δεν μπορεί να ε, υπάρξει χωρίς τη συγκατάθεση των κρατών μελών γιατί δεν είναι ε, αναλογικό μέτρο. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κάποιον κανόνα, κάποια νομοθεσία σχετικά με την προσφυγή σε, κράτος, σε δικαστήριο κράτους μέλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. Ε, η κυρία Μινέρα έχει το λόγο πρώτη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Χίντελαν για αυτή την εξαιρετική και πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ε, τη δεν ε, την έχω καταλάβει ε, απόλυτα, πρέπει να ομολογήσω. Γι' αυτό έχω αρκετές ερωτήσεις. Μας είπατε πώς πρέπει να γίνει μία ε, αλλαγή. Μας μιλήσατε για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ, μας μιλήσατε για επιστροφή σε ε, εθνικά ε, δικαστήρια. Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή. Αυτή η αλλαγή οφείλεται σε άλλους λόγους πέραν της αρχής της επικουρικότητας. Μετά, η διαιτησία. Ένας τέτοιος διαιτητής θα μπορούσε να ε, ασχολείται με πολλές υποθέσεις ταυτόχρονα. Αυτό απαγορεύεται, θα έπρεπε να απαγορεύεται. Υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Και ε, τρίτον, οι αποζημιώσεις ε, είναι κάτι που δεν αποφασίζει η Επιτροπή. Υπάρχει μια διρυθμιστική αρχή όπου οι επενδυτές απειλούν με προσφυγή για να μην υπάρξει αυτή η για να μην, μπορούν, να, μην χρειαστεί να πληρώσουν αποζημίωση. Τι γίνεται, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί. Μετά, ο μηχανισμό ιδιαιτησίας στην συμφωνία ΣΕΤΑ και στη συμφωνία με το Βιετνάμ ε, έχουν αρκετά προβλήματα. Ε, υπάρχει όμως κάποιος μηχανισμός διαιτησίας ο οποίος να είναι πιο οικονομικός, πιο προσεκτός, πιο εύκολος ή η διαιτησία είναι πάντα η ακριβότερη λύση και ποιε είναι οι προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε εκείνη να ε, προβεί σε λύσεις. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα ήθελαν το λόγο. Εάν όχι, θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση. Ε, να πω πρώτα ότι και εγώ τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συγκαπούρης την καταλαβαίνω ε, ως εξή Υπάρχουν κάποιοι κανόνες ε, που σύμφωνα με αυτούς πρώτα πρέπει να εξαντληθούν οι εθνικές δυνατότητες στα προσοχή στα δικαστήρια κτλ. Και μετά να περάσει το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην αρμοδιότητά της. Έτσι καταλαβαίνω τουλάχιστον την μεικτή αρμοδιότητα έτσι όπως αναγράφεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μετά υπάρχουν αυτές οι επενδύσεις χαρτοφυλακίων, portfolio investment. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Εδώ υπάρχει δυνατότητα να έχουμε μία σαφή ε, πολιτική, μια σαφή κατεύθυνση έτσι ώστε να μην ε, έτσι επιλύονται αυτές οι διαφορές. Τώρα υπάρχουν οι πολυμερείς συμφωνίες και εκεί τι γίνεται, ποιο δικαστήριο θα δεχτεί να αναλάβει μια τέτοια υπόθεση, από ποιους δικαστές θα αποτελείται, τι σύνθεση θα έχει. Ε, ιδιαίτερα στην περίπτωση πολυμερών συμφωνιών όπου κάποιοι εταίροι δεν ανήκουν στις ε, ανεπτυγμένες χώρες. Ε, είναι... Ποια θα είναι λοιπόν η σύσταση αυτού του δικαστηρίου και αυτό το δικαστήριο με την όποια σύνθεση θα γίνει αποδεκτό από όλους τους εταίρους. Υπάρχουν θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία δείχνουν ε, ελλειπή ανοχή. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, θα, εμπορε, θα μπορούσε να υπάρξει ένα διεθνές επενδυτικό δικαστήριο το οποίο θα προβλέπει δράση και αυτές τις περιπτώσεις. Μετά, μετά από όλα αυτά θα δώσω, πίσω το λόγο, θα δώσω μάλλον το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Αντρέφον Βάλτερ, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει με αυτήν την πρόταση για Διεθνές Επενδυτικό Δικαστήριο. Μετά θα ήθελα να ρωτήσω επίσης και λεπτομέρειες σχετικά με την εκτίμηση αντικτύπου που έχει διεξαχθεί και ε, θα με ενδιαφέρει πολύ να μάθω τα αποτελέσματα της μελέτης. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω το λόγο στον κύριο Φων Βάλτερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον καθηγητή Χίντελεν για την παρουσίασή του και τα αποτελέσματα της μελέτης. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να αντιδράσω στην παρουσίαση του κυρίου Χίντελεν και μετά θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Κάρλο, ο οποίος θα σας παρουσιάσει μια συνοπτική εικόνα της ε, επενδυτικής μας πολιτικής και το τι συμβαίνει με αυτό το Διεθνές Επενδυτικό Δικαστήριο. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσω πολύ σύντομα και να σχολιάσω αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Με μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν άκουσα αυτά που μας είπατε. Πιστεύω πως είναι πολύ επίκαιρη αυτή η μελέτη ακριβώς επειδή προσπαθούμε να δούμε τις λεπτομέρειες στο project αυτό του δημιουργία Διεθνούς Επενδυτικού Δικαστηρίου. Να δούμε δηλαδή ε, όχι μόνο ε, το πλαίσιο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και από άλλα ε, παγκόσμια όργανα διαιτησίας διαμεσολάβησης έτσι ώστε συνδυάζοντας τις διάφορες πτυχές τους να βρούμε την ε, βέλτιστη δυνατή λύση. Θα ήθελα λοιπόν πολύ σύντομα να κάνω τα εξής σύντομα σχόλια σε αυτά που άκουσα. Σε ό,τι αφορά βέβαια τις ειδικές μας διαπραγματεύσεις που ολοκληρώθηκαν. Το πρώτο λοιπόν σχόλιο έχει ως εξή. Νομίζω πως όλοι γνωρίζετε αυτά που λέγονται για την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συγκαπούρης, για το τι μπορεί να γίνει και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την συμφωνία έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούμε με τις αντίστοιχε ε, συμφωνίες ΣΥΤΑ και τη συμφωνία με το Βιετνάμ, να ευθυγραμμίσουμε το κείμενο. Υπάρχουν ορισμένα σημεία της Συμφωνίας ΣΥΤΑ και της Συμφωνίας με το Βιετνάμ όπου αναφέρεται η παραδοσιακή διαιτησία όπως ε, αναφέρεται και στις διάφορες συνθήκες. Θα μου επιτρέψετε εδώ να διαφωνήσω σχετικά με το τι καθιστά μια διαιτησία παραδοσιακού τύπου. Η μελέτη δηλαδή αναφέρει ότι πρέπει να συνεχίσουμε, να διατηρήσουμε το status quo να, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διατησία. Αυτό είναι κάτι όμως που πρέπει πρώτα να συζητηθεί με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε λύσεις. Δεν πρέπει να αφαιρείται η αρμοδιότητα των κρατών μελών εδώ να αποφασίσουν. Και μετά, υπάρχει και η ανάλυση του τι καθιστά τυπική παραδοσιακή ε, διαιτησία σε διαφωνίες επενδυτών και κράτους. Ε, το θέμα εδώ νομίζω πως ε, είναι το εξής. Ε, πρέπει να δούμε πόση μεταρρύθμιση σηκώνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γιατί υπάρχουν πολλέ προκλήσει, υπάρχουν πολλά θέματα και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί από τη μελέτη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε αυτό που προχωρήσουμε σε, πολυμερές, σε πλαίσιο. Μετά υπάρχουν και κάποια Κάποιε μικρέ λεπτομέρειε ε, που με βρίσκουν αντίθετο στη μελέτη. Για παράδειγμα υπάρχει η δήλωση ότι στη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη δεν υπάρχουν κάποιε ρήτρε για, για την εφαρμογή των διατάξεων. Μετά υπάρχουν κάποιε αναφορέ σε μελέτες, αλλά θα ήθελα πρώτα να υπάρχουν αυτέ οι μελέτε και μετά. Αυτά λοιπόν προ το παρόν. Επιτρέψτε μου να σταματήσω εδώ και να δώσω το λόγο στον ε, Κάριλ, ο οποίο θα σα δώσει μια συνοπτική εικόνα του πλαισίου για το Διεθνέ Επενδυτικό Δικαστήριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε λοιπόν στο state of play της επενδυτικής πολιτικής. Σωστά. Ναι. Ωραία. Ας δώσουμε πρώτα λοιπόν το λόγο στον ε, κύριο Χίντελανγκ να απαντήσει θα έλεγα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να πω. Καταρχάς ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Μετά, γιατί χρειαζόμαστε αυτήν την, ε, την ε, διαιτησία επενδυτών κράτους της στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Συμφωνιών. Πιστεύω ότι καταρχάς όλοι έχουν υπογράψει τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μετά, ναι, μπορεί να υπάρξει ε, προκατάληψη ε, απέναντι σε έναν ξένο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αποφευχθεί αυτό. Αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από την ε, διαιτησία επενδυτή και κράτου. Πρωτού κλείσουμε λοιπόν αυτά τα κεφάλαια. Τώρα γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσία ε, έχουν τόσο μεγάλη δυσκολία πρόσβασης. Καταρχάς, αναφέρθηκε ότι το μέσο κόστος προσφυγής σε διαιτησία ήταν πριν από κάποια χρόνια 8 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα έχει ανέβει στα 12 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το χρήμα είναι στο κέντρο. Το χρήμα εμποδίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε διαιτησία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε ε, ευφυείς, να βρούμε καλές λύσεις, να δουλέψουμε με άλλα ε, με άλλες πιθανότητες πρώτου προσφύγουμε σε διατησία, έτσι ώστε να ωφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κύριο όμως ε, μέλημα μας πρέπει να είναι, να είναι δικαστήρια, εθνικά δικαστήρια που θα είναι αποτελεσματικά. Τώρα, σχετικά με την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την συμφωνία με τη Σιγκαπούρη, να πω ότι πράγματι Τα ευρήματα του δικαστηρίου στην επίλυση διαφορών επενδυτή και κράτους ε, είναι, έχουν ως εξή. Δεν χρειάζεται να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες ε, πριν. Αλλά μπορούμε καταρχάς να χρησιμοποιήσουμε τα εγχώρια ένδικα, ένδικα μέσα, να προσφύγουμε στο Εθνικό Δικαστήριο. Τώρα, ε, εάν υπάρχει μεικτή αρμοδιότητα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκήσει αυτό το δικαίωμα, τότε τα κράτη-μέλη θα μείνουν εκτός διαδικασίας. Τώρα στα, στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, εδώ δεν ε, πιστεύω υπάρχει λόγος ανησυχίας, εφόσον υπάρχει πολιτική θέληση για να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Όμως το δικαστήριο εδώ δεν ήταν σαφές και θα περιμένουμε λοιπόν ε, και συνέχεια περισσότερες ε, έρευνες. Τώρα, πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο. Ναι, αυτό θα ήταν πολύ λογικότερο. Ε, το οποίο θα αντικαθιστούσε και όλα στις ε, μεγάλες, μακρές διαδικασίες επίλυσης διαφορών με διμερείς συμφωνίες. Όμως, μην ξεχνάτε ότι αυτό συνεπάγεται και πρώτερες συμφωνίες, συνεπάγεται κάποια κοινά ουσιαστικά πρότυπα και εδώ θέλω να ευχηθώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλή τύχη γιατί είναι μεγάλο το κουβάρι. Υπάρχουν κάποια ιστορικά ε, πλαίσια όπως η Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η οποία ε, όμως προσθέθηκε αργότερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λέγκ. Πάντα μας είναι πολύ ευχάριστο όταν έρχεστε και μας παρουσιάζετε τις μελέτες σας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ και προσμένουμε σε συνέχεια της συνεργασίας μας. Τώρα λοιπόν θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 5-6 λεπτά, έτσι ώστε να μας ενημερώσει για τις νεότερες εξελίξεις και το τι σκέφτεται η Κομισιόν για την επενδυτική πολιτική. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. αφού έχω το χρόνο να σας πω πώς έχουν τα πράγματα για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά εμείς σας τα πω όλα, θα πρέπει πάρα πολύ χρόνο. Μόνο τρία θεματάκια πρώτα πρώτα όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού BIT και τι γίνεται με το Διεθνές Δικαστήριο Επενδύσεων και τι γίνεται με τη νέα ανακοίνωση. Πρώτα πρώτα. Από τότε που ετέθησε η ισχύ αυτός ο κανονισμός serves the management of the existing bilateral investment treaties of member states and the authorization of new bilateral investment treaties. Για αυτές τις συμφωνίες, τις διμερείς για τις επενδύσεις. Πρόκειται για την ρήτρα δικαιωμάτων. Όσον αφορά τις υπάρχουσες συμφωνίες, έχουμε δηλαδή 24 αποφάσεις για να υπογράψουν 19 νέες συμφωνίες στα κράτη-μέλη και 21 πρωτόκολλα και 24 αποφάσεις που εγκρίνουν τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν ενισχύ 16 συνθήκες που υπογράψαν μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και 17 πρωτόκολλα που προηγήθηκαν. Όλα αυτά βέβαια σε κάποια στιγμή ανεστάλησαν γιατί είχαμε με τις εγκρίσεις αυτές για άλλες ε, διαπραγματεύσεις, γιατί είπαμε το θεματολόγιο από το Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιούνιο του 2016 να, ε, να θεωρηθεί, οπότε δεν δώσαμε άλλες εγκρίσεις, γιατί ήμασταν στη διαδικασία της μεταρρύθμισης. Οι κανόνες, οι κανόνες θέσπισης ε, νομοθετημάτων και το νέο σύστημα επίλυσης διαφόρων. Οπότε κάτι αν θέλουν, μπορούν να κάνουν διαπραγματεύσει. Αλλά πρώτα-πρώτα θα πρέπει να φυλαμίζονται με τι διατάξει του ειδικού δικαίου και θα πρέπει επίση να συμβαδίζουν με τη νέα μα προσέγγιση για τι επενδύσει. Και έτσι όλοι να κινούμεθα στην ίδια κατεύθυνση. Και γι' αυτό έχουμε κάποιε συγκρίσει που εκκρεμούν. Δεν προέβημε σε αυτέ, διότι σε κάποιες περιπτώσεις τα κρατημέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν τον πρότυπό στη νέα προσέγγιση και δεν το είχαν πράξει. Επίσης, κάποιες άλλες ε, ειδοποίησεις για σύννεψη συμφωνίων γιατί δεν υπήρχε πλήρης ευθυγράμμιση ακόμη με το γενικό δίκαιο, οπότε γι' αυτό και ακόμη είμαστε στη φάση της συνεννόησης. Επίσης, ε, είπαμε για διατήρηση σε ισχύ κάποιων συμφωνιών αλλά σε περιπτώσεις που υπήρχαν κάποιες ασυμβατώσεις με το κοινωτικό δίκαιο. Άρα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιλύσουμε τα σχετικά προβλήματα. Κάποιες από αυτές τις ε, εγκρίσεις αφορούν κάποιες συνθήκες που θεωρήθηκαν ασύμβατες με το κοινωτικό δίκαιο λόγω της transfer clause, γιατί δεν είχαν τις σχετικές ρήτρες διαφύλαξης και είχε κρίνει το δικαστήριο ότι υπάρχει ασυμβατότητα για αυτές τις ρήτρες οπότε είπαμε στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να προσαρμόσουν αυτέ τι ρήτρε στο κοινοτικό δίκαιο. Από ό,τι θα θυμάστε, οφείλαμε να αναφέρουμε σχετικά σε Συμβουλή και Κοινοβούλιο για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 όμως η σχετική έκθεση θα υποβληθεί σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο μέσα στο 2018 και εκεί θα αναφέρουμε τα της εφαρμογής του κανονισμού. Και αν χρειαστεί θα υπάρξουν και αλλαγές. Τώρα όσον αφορά αυτό το πολυεθνικό, διεθνές τέλο πάντων δικαστήριο επενδύσεων. Είχαμε ένα ιντερνετικό ερωτηματολόγιο, οπότε μας απήντησαν 193, λάβουμε 45 επίση έγγραφα από συνδικάτα, από τη βιομηχανία, από πανεπιστήμια κλπ. Όλες οι απαντήσεις υπάρχουν στο website. Και έτσι όλα αυτά θα μπουν σε κάποια έκθεση που θα είναι έτοιμη όταν ε, η τελική αξιολόγηση θα είναι έτοιμη. Αλλά όλα αυτά θα τα απαντήσουν πρώτα στο website. Το αποτέλεσμα αυτής της διαβουλεύσης που κάναμε δείχνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι υπέρ αυτή της πρόταση για ένα διεθνέ δικαστήριο επενδύσεων. Και επομένω, όλοι συμφωνούν. Χρειάζεται ένα τέτοιο δικαστήριο. Ο καθένας βέβαια έχει σε επιμέρου ζητήματα διαφορετικές απόψεις. Οπότε τον Ιούλιο θα παρουσιάσουμε το σχέδιο της ε, μελέτης αξιολόγηση, οι επίτροποι θα συζητήσουν την διαπραγματευτική εντολή περί τα τέλη του 2017 και όλα αυτά θα παρουσιαστούν μαζί με την έκθεση της μελέτης επιπτώσεων. Θα ως δεύτερο σημείο το Διεθνές Δικαστήριο ε, των επενδύσεων, τρίτο σημείο. Ο απολυναντισμός μας όσον αφορά αυτή τη νέα ανακοίνωση στην ε, ανακοίνωση για το εμπόριο για όλους είπε μας θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με την ανακοίνωση του 2010 οπότε και του χρόνου θα επικαιροποιήσουμε τα σχετικά όταν θα αναζητήσουμε νέους τρόπους ε, για το πώς θα χαράξουμε την επενδυτική μας πολιτική Είμαστε στη φάση τώρα της ε, ολοκλήρωσης, της τελικής φάσης, ώστε να ξεκινήσουν όλα αυτά. Οπότε και το δεύτερο εμείς του 2017 θα έχουμε διαβούλευση για όλους τους εμπλεκομένους και έτσι θα γίνουν επαφές, συζητήσεις και στο Κοινοβούλιο με τους εμπλεκόμενους και θα συνταχθεί αυτή η νέα ανακοίνωση του 2018 η οποία και θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο του 2018. Αυτά και ευχαριστώ. So, September 18. Ευχαριστώ πολύ. 18 ε, λοιπόν Σεπτεμβρίου, ελπίζω να μπορέσετε να είστε εκεί, γιατί η θητεία μας λύγει το Μάιο του 2019. Ελπίζω λοιπόν να είμαστε γρήγοροι και να πιέσετε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ όλους. Εδώ ολοκληρώνεται το δημόσιο κομμάτι της συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Θα αρχίσουμε αμέσως την ε, συνεδρίαση των συντονιστών η οποία θα γίνει και κλεισμένον των θυρών. Έχετε λοιπόν ένα λεπτό να εγκαταλείψετε την αίθουσα.